Präsident! Vielen Dank. Guten Tag, meine. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσετε τις θέσεις σας. am 19. Januar Ιανουαρίου 2012 διακόπη συνεδρίαση η οποία τώρα συνεχίζεται τα πρακτικά της συνεδρίας της 19ης Ιανουαρίου 2012 και τα εν λόγω κείμενα είναι ενώπιόν σας. Υπάρχουν διαφωνίες, παρατηρήσεις. Όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά αυτά. Πέραμε σε ανακοινώσει του Πρόεδρου. Δύο βουλευτέ δήλωσαν ότι <coughs> κρατούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρια νταιαννα Νταγιάννα Βόλη. Από 1η Φεβρουαρίου 2012 γράψει στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βόλης για την πολυετή επικοδομητική και επιτυχή εργασία της για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, ο κ. Πρόεδρος Αστερόσα ανακοίνωσε ότι από την Δευτέρα Φεβρουαρίου καταθέτει την εντολή του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τα συγχαρητήρια εσύ και για τον ίδιο. Ελπίζω ότι θα έρθει σε λίγο και μπορείς να το ευχαριστήσω και προσωπικά. Το σώμα το σημειώνει και η βάση του άρθρου 4, παραγραφή 1 και 3 του κανονισμού, σημειώνει ότι οι έντρες αυτές χειρεύουν από τις ημερομηνίες που προανέφερα. Ο κ. Ιταλά μου ανακοίνωσε ότι ορίστηκε μέρο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Το σημειώνει το Κοινοβούλιο αυτό και βάσει το άρθρο 4, παραγράφη 1 και 4 του κανονισμού σημειώνει την χειρία τη έδρα του κ. Βίταρ Ιταλά από την 1η Μαρτίου 2012. Θα ήθελα επίση να σα ανακοινώσω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Συνεδρία τη 25 Ιανουαρίου τρέχοντο έτου, έλεγξε μια σειρά εντολών βάσει του κανονισμού άρθρο 3, παράγραφος 3 και 4 και προτείνει τους εξής. Ε, Άντερ Στότερ, Κουσκέρι, Γκαρσία Ραμόν, Γκαρσία Ιέρο Καραβάλο, Μακίνταερ, Μαλινόφ, Νίλσον, Ότις Βιλέλα, Σαρτούρσκι, Σέντο Ιαλαμπάρ, Τρεματέρα και Βάρνχολτσα. Μπρατκόφση, Κοσέ Ροάτα Στάντλερ, Κούκοβιρ, Φαντεστούφ, Μιράνο Μάριε, Κορέα Ζαμόρα, Ναράχο Εσκομπάρ και Σούμπερ. Είναι κανείς κατά του ορισμού των μελών αυτών. Όχι, οπότε ε, επικυρώνεται η έγκριση. Από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού του ε, των Σοσιαλιστών, των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και την ΓΚΟΕ, Έχω μια σειρά αιτούσεων για ορισμό μελών σε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και αντιπροσωπείε. Ο ελόγω κατάλογο θα ε, παρατηθεί στα πρακτικά τη τρέχουσα συνεδρίαση. Αν μέχρι την έγκριση των πρακτικών δεν υπάρχει διαφωνία, ισχύουν αυτοί οι ορισμοί. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων επίση προτείνει την εξή διόρθωση ενό από τα κείμενα τα οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Για τον κορισμό 596 κάθε 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή κάποιων νομικών πράξεων στην διακανονιστική διαδικασία. Με έλεγχο. Τέταρτο τμήμα. Και υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος γράφων κομισιών, συμβουλίου κλπ. Δεν πρόκειται να σας τον διαβάσω τώρα. Θα μπορείτε να το δείτε άμεσα στο Sion Direct και έτσι θα κάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου. Περνάμε τώρα στο πρόγραμμα εργασίας, στο οριστικό και η πρόταση του ημερησίας διάταξης αποθετήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του Προέδρου, στις 19 Ιανουαρίου του διάσκεψη του Προέδρου. Θέλω κάποιο από αυτό το λόγο. Όχι. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω. Η συζήτηση για τα συμπεράσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 30 Ιανουαρίου 2012 θα λάβει τώρα από τις 3 και 10 έως τις 5 παρά 20 χώρα. Η ώρα των ερωτήσεων προς την είπα το εκπρόσωπο θα γίνει 5 παρά 20 έως 6 ε, παρά 20 και οι επόμενε συζητήσει θα αρχίσουν στις 6 παρά 20. Η συζήτηση για την έκθεση του Ουργαΐζα Αγγουλό για την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα θα αναβληθεί μέχρι την Πέμπτη. Η επερώτηση για την προφορική ερώτηση για την εφαρμοσιμότητα της, ε, ε, των, ε, των, των, των ομολόγων σταθερότητα θα ανεκατασταθεί από την Τουρβάζη Άγκολο. Επίσης, θα έχουμε μια συνομή παρουσία τη έκθεση ΡΕΚΒΑ και η πρόταση ψηφίσματος για την ε, προσθέμενη αξία που προσθέτει ε, προτείνει το, η Επιτροπή Περιβάλλοντος σύμφωνα με το 88 κάθετος 2 θα περάσει αμέσως στην ψηφοφορία. Αν διαφωνεί κανένας, όχι βλέπω όλοι ενθουσιώδης υπέρ, αποφασίζεται αυτό. Και τροποποιείται έτσι η ημερησία διάταξη. Περνάμε τώρα στις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα συμπεράσματα του τύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30 Ιανουαρίου 2012. Και χαιρετίζω από αυτού τον κύριο Ρομπόη, πρόεδρο της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον κύριο Μπαρόζο, πρόεδρο της Επιτροπής και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο κύριο Ρομπόη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία δύο χρόνια οι Ευρωπαίοι ηγέτες έπρεπε να πάρουν δύσκολες και συχνά επώδυνα μέτρα για να σταθεροποιήσουν την Ευρωζώνη. Παρότι αυτό ήταν αναγκαίο και τώρα